Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά λοιπόν της 7ης ε, Ιουλίου είναι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω κατά αυτόν. Έχουν εκριθεί λοιπόν τα πρακτικά.